Εδώ η ψήφιση θα διαξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου τον Ιούνιο. Η επόμενη συνεδρίασή μας στην Ολομέλεια θα είναι αύριο Τετάρτη 22 Μαΐου στις 8.30 το πρωί. Πρώτο τμήμα μέχρι τις 14.00 και το δεύτερο τμήμα από 15.00 έως